deschisă ședința de astăzi. Primul punct pe ordinea de zi. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η συνεδρίαση. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Συζητήσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και